για την νομοποίηση εσόδων παράνομες δραστηριότητες της χρηματοδότησης τρομοκρατίας και που τροποποιεί την οδηγία του 2009 κάθετο 109 έχει ως στόχο να βελτιώσει την πρόσφατη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τη χρηματοπιστωτική διαφάνεια και τους χρηματοπιστωτικούς ελέγχους προκειμένου να αυξηθεί η καταπολέμηση της νομοποίησης ε, εσόδων παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότης τρομοκρατία. Έχουμε τα εξή βασικά προβλήματα. Πρώτον, οι ύποπτε συναλλαγέ που αφορούν τρίτε χώρε υψηλού κινδύνου δεν παρακολουθούνται αποτελεσματικά λόγω των ασαφών και μη συντονισμένων απαιτήσεων για τη διενέργεια δέουσα επιμέλεια ω προ τον πελάτη. Δεύτερον, έχουμε ύποπτε συναλλαγέ με τη χρήση εικονικών νομισμάτων που δεν παρακολουθούνται παρκώς από τι αρχέ, οι οποίες τελικά δεν είναι καν σε θέση να κάνουν τη σύνδεση ταυτοτήτων και συναλλαγών. Τρίτον, τα εφιστάμενα μέτρα για τον περιορισμό των κινδύνων νομοποίηση εσόδων παράνομη δραστηριότητα ή χρηματοδότηση τρομοκρατία που συνδέονται με τα νόμιμα προπληρωμένα μέσα είναι ανεπαρκή. Τέταρτον, οι μονάδε χρηματοοικονομικών πληροφοριών δεν έχουν πρόσβαση και δεν ανταλλάσσουν πληροφορίε που κατέχουν οι υπόχρεε οντότητε. Πέμπτον, οι μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών στερούνται πρόσβαση ή έχουν καθυστερημένη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα των κατόχων τραπεζικών λογαριασμών και λογαριασμών πληρωμών. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να βρεθεί σωστή ισορροπία ανάμεσα στη θέσπιση επαρκών ελέγχων για την αποτελεσματική αποτροπή των οικονομικών εγκλημάτων και της χρηματοδότης τρομοκρατίας, αφενός και στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και των θεμελιωδών δικαιωμάτων αφετέρου. Χρειάζονται ξεκάθαροι κανόνες που θα μπορούν πραγματικά να δυναμώσουν την παρακολούθηση από τράπεζες, λογιστές και όλους τους υπόλοιπους επαγγελματίε του τομέα. Βάσει λοιπόν και της πρότασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών θα μπορούσαν να ελέγχουν τις διευθύνσεις που χρησιμοποιούν οι κάτοχοι οικονομικών νομισμάτων. Επίσης, η χρήση των ανώνυμων προπληρωμένων μέσων και καρτών, χωρίς να έχει γίνει ο έλεγχος δέουσας επιμέλειας, θα πρέπει να μειωθεί και θα πρέπει το επίπεδο να είναι τα 150 πλέον ευρώ, ενώ θα πρέπει να μην επιτρέπονται οι υπόλοιπε πληρωμές. Βέβαια, οι περιορισμοί αυτοί δεν θα πρέπει να είναι τόσο αυστηροί, που να καταστήσουν τελικά τις κάρτες αυτές άχρηστες στην πράξη. Επίσης νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχουν κεντρικά μητρώα αρχεία για τους α, κατόχους τραπεζικών λογαριασμών. Επίσης θα πρέπει να δίδεται στις αρμόδιες αρχές πρόσβαση όσον στα μητρώα εκείνα όπου βλέπουμε πραγματικά ποιοι είναι οι δικαιούχοι και οι διοκτήτες συγκεκριμένων καταπιστευματικών εταιριών και επίσης θα πρέπει να παρακολουθούμε ακόμα περισσότερο τις συναλλαγές με τις τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου. Επομένως, οι τρεις βασικές γραμμές της πρώτας Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρέπει να στηριχθούν με κάποιες όμως τροπολογίες που έχουν ως στόχο να ενισχύσουν την καταπολέμηση της νομοποίησης εσόδων παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότης τρομοκρατίας με παράλληλη διασφάλιση του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε αυτό το πεδίο σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να υπάρχουν κενά στην νομοθεσία τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν οι κλιματικέ οργανώσει. Το εφιστάμενο χρηματοπιστωτικό σύστημα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για να ξεπλένονται τα χρήματα τη μαφία ή να χρηματοδοτείται η τρομοκρατία. Τα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και οι εθνικέ αρχέ θα πρέπει να καταβάλουν περισσότερε προσπάθειε προκειμένου να αντιμετωπίσουν το πολύ σημαντικό αυτό ζήτημα. 12 Δεκεμβρίου του 2016 είναι μάλιστα και προθεσμία υποβολή τροπολογιών, λέει ο εισηγητής. Στι σημειώσει μου λέει 8 Δεκεμβρίου. Ας το δούμε. 8 λοιπόν Δεκεμβρίου είναι η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών. Κύριε Ράντιεφ, θέλετε να πάρετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Σα όδης ε, εισηγητής. Ε, θα ήθελα και εγώ να κάνω κάποιες προτάσεις, οι οποίες ουσιαστικά ακολουθούν το γενικό προσανατολισμό του ε, σχεδίου έκθεσης το οποίο θα συζητήσουμε σε κοινή συνευρίαση της ΛΥΠΕ και της ΕΚΟΝ την Πέμπτη. Θα υποβάλουμε κάποιες τροπολογίες, δεν μπορώ να σας τις οριστικοποιήσω τώρα, καθότι δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα οι τροπολογίες αυτές. Πάντως είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε μια πολύ επικοδομητική συνεργασία. Αυτό που θέλουμε είναι σε κάθε περίπτωση να προχωρήσουμε σε ένα σύστημα πρόληψης, τη νομοποίηση εσόδων παράνομε δραστηριότητε, θέλουμε προφανώ να πατάξουμε τη χρηματοδότηση τη τρομοκρατία. Αυτό το οφείλουμε στου Ευρωπαίου πολίτε. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελε η Κομισιόν να τοποθετηθεί. Όχι. Αυτά λοιπόν για το θέμα αυτό. Παρότι έχουμε αναβάλει τη συζήτηση του σημείου 7, επί τα αποέτοιμα του κ. Λεμπρετών, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών είναι η 9η Δεκεμβρίου. Περνάμε στο θέμα 8, εξέταση σχεδίου γνωμοδότησης για την τροποποίηση της οδηγίας 2004 κάθετος 37 και σε αυτή την περίπτωση συντάξεις γνωμοδότησης είναι ο κύριος Χρυσόγονος. Ευχαριστώ κύριε ε, Πρόεδρε. Ο καρκίνος στην εργασία είναι ο υπαριθμόν ένα λόγος θανάτου στον ε, αναπτυγμένο κόσμο και η πολύ σοβαρή αυτή ασθένεια ε, καθίσταται ο σημαντικότερος λόγος θανάτου. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμάται ότι άνω των 100.000 θανάτων ε, ε, οφείλονται κάθε χρόνο σε καρκίνο ε, που προκαλείται από την εργασία. 50.000 νέα περιστατικά εμφανίζονται κάθε χρόνο. Ο καρκίνος λοιπόν είναι ο υπαριθμόν ένα λόγος θανάτου στην Ευρωπαϊκή Ένωση για επαγγελματικούς λόγους, ανερχόμενος στο 53% των θανάτων. Περίπου 20 εκατομμύρια εργαζόμενοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκτίθενται σε καρκινογόνες ουσίες. Ο θάνατος από τον καρκίνο, ο καρκίνος μάλλον, οφείλ, ε, ευθύνεται και για μείωση της ποιότητας ζωής, αλλά και για ε, δαπάνες για τα κοινωνικά συστήματα. Επίσης, ο καρκίνος ε, επηρεάζει την οικονομική ευημερία καθώς αναγκάζει ε, τα κράτη να καταβάλουν επιδόματα και να χρηματοδοτούν τα συστήματα ιατρικής περίθαλψης. Επίσης, ευθύνεται για την απώλεια παραγωγικότητας, καθώς και για την ε, υποχρέωση ε, καταβολής υψηλότερων μισθών λόγω ε, υψηλότερου κινδύνου κατά τη ζωή, κατά την εργασία. Η πρόταση για την τροποποίηση της οδηγίας 2004-37 σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνου παράγοντες που συνοδεύεται από μελέτη αντικτύπου έχει ως στόχο την προστασία των Ευρωπαίων εργαζομένων μέσω της θέσπιση υψηλότερων προδιαγραφών σε ενωσιακό επίπεδο προστατεύω του εργαζομένους από την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες. Η σκοπή της πρότασης είναι να ε, ενισχυθεί και να βελτιωθεί η προστασία της υγείας από την ε, έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες, να εξασφαλίσει σαφήνεια και να δημιουργήσει καλύτερους όρους ανταγωνισμούς για τους οικονομικούς φορείς και τρίτον να αυξήσει την αποτελεσματικότητα του ευρωπαϊκού πλαισίου για την προστασία των εργαζομένων επικαιροποιώντας το στη βάση των ε, διαθέσιμων επιστημονικών στοιχείων. Οι στόχοι αυτοί ε, είναι συνεπής με το θεμελιώδες δικαίωμα στη ζωή και σε δίκες συνθήκες εργασίας με το σεβασμό της ανθρώπινης ζωής ε, και αξιοπρέπειας όπως προβλέπεται και στην Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σκοπός της πρότασης είναι να εντάξει στην νομοθεσία μια σειρά από χημικές ουσίες που έχουν αναγνωριστεί ως καρκινογόνες σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από διεθνείς οργανισμούς όπως είναι ο το Διεθνές Συμβούλιο για την Έρευνα για τον Καρκίνο, αλλά δεν ταξινομούνται ακόμα βάσει του ισχύοντος ευρωπαϊκού πλαισίου. Συγκεκριμένα, προτείνει να αναθεωρήσει τη, τα όρια ε, ε σε ε, ε, επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για 13 παράγοντες στη βάση των τελευταίων επιστημονικών ενδείξεων εναρμονίζοντας με αυτόν τον τρόπο τα διάφορα εθνικά όρια όπου αυτά υπάρχουν. Αυτό εκτιμάται ότι θα, θα διασώσει 100.000 ε, ε, ανθρώπινες ζωές έως το 2020 ε, ε, και θα εξοικονομήσει έως 90 δισεκατομμύρια ευρώ. Γι' αυτό το λόγο υποστηρίζω με ορισμένες τροπολογίες βέβαια την πρόταση που οι τροπολογίες μου αφορούν κυρίως την προσέγγιση προφύλαξης που θα πρέπει να ενισχυθεί στην πρόταση αυτή. Η, τα όρια λοιπόν για αυτές τις καρκινογόνες και μετακληρογόνες ουσίες θα πρέπει να αναθεωρούνται τακτικά βάσει των ε, επιστημονικών ενδείξεων καθώς και βάσει των τεχνολογικών εξελίξεων όσον αφορά την μέτρηση και την πρόληψη κινδύνων η αρχή της προφύλαξης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ε, σε γενικό επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία προκειμένου να εξασφαλιστεί η προστασία των καταναλωτών, των εργαζομένων και του περιβάλλοντος σε όλους τους τομείς δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνιστάται λοιπόν εκεί όπου υπάρχουν ανεπαρκείς ή ανολοκλήρωτες επιστημονικές ενδείξεις και όπου υπάρχουν ενδείξεις ότι ενδεχόμενες επιπτώσεις στο περιβάλλον, την υγεία των ανθρώπων, των, των ζώων ή των φυτών, θα πρέπει να ε, ακολουθείτε πάντοτε ένα υψηλό επίπεδο προστασίας. Αυτό πρέπει να ε, ακολουθηθεί και στην περίπτωση ε, των ε, τοξικών μειγμάτων και των επιπτώσεών τους στην υγεία των εργαζομένων. Αυτό είναι απαραίτητο προκειμένου να επιτευχθεί μια αποτελεσματική ε, πρόληψη του καρκίνου η οποία θα λαμβάνει υπόψη όλα τα επιστημονικά και τεχνολογικά δεδομένα της εποχής μας. Πρέπει να σημειωθεί ότι προκειμένου να προστατευτούν οι εργαζόμενοι από τους κινδύνους που προκαλούνται από την έκθεσή τους σε καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους παράγοντες υπάρχουν μια σειρά από ουσίες οι οποίες ακόμη δεν εντάσσονται στην ε, πρόταση αλλά ταυτόχρονα θα μπορούσαν να επηρεάσουν και να πλήξουν την υγεία των εργαζομένων. Όλες οι ουσίες που ενδέχεται να είναι καρκινογόνες θα πρέπει να καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία προκειμένου να εξασφαλίζονται ε, οι συνθήκες ζωής, διαβίωσης, υγείας όλων των Ευρωπαίων πολιτών. Η Ευρωπαϊκή πρέπει να, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να καταβάλει σοβαρότατες προσπάθειες προς αυτόν τον στόχο και θα πρέπει να ε, υποβάλει ένα πρόγραμμα για την εξάλληψη του καρκίνου λόγω έκθεσης κατά την εργασία. Σε συνεργασία με το Διεθνές Γραφείο Εργασίας και τον ΟΗΕ ε, πρέπει να ε, υπάρξει, να συνταχθεί και να εκπονηθεί ένα τέτοιο πρόγραμμα. Ταυτόχρονα θα πρέπει να εκπονηθεί και μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο στην εργασία. Τέλος, ε, στις διαδικασίες θα πρέπει να ακολουθούν διαδικασίες περιορισμού των καρκινογόνων μεταλλαξιογόνων παραγόντων όπου αυτό είναι δυνατόν. Ε, κυρία Ρέγνα έπρεπε να φύγει, έπρεπε να πάρει την κόρη στο σχολείο, να πάρει την κόρη από το σχολείο. Μου ζήτησε λοιπόν να διαβάσω την δήλωσή της. Υποστηρίζω τόσο την θέση του συντάκτη της γνωμοδότης όσο και την πρόταση της Κομισιόν. Εμείς εδώ και πάρα πολλά χρόνια υποστηρίζουμε την βελτίωση του συστήματος προστασίας των εργαζομένων στον χώρο εργασίας τα προστατευτικά μέτρα για την υγεία των εργαζομένων θα πρέπει να εφαρμόζονται προτού ασθενήσουν οι εργαζόμενοι. Αυτό αφορά και τον χρόνο εργασίας αλλά και τον χρόνο μετά την ολοκλήρωση της ε, εργάσιμης ζωής του πολίτη. Γιατί ε, οι επιπτώσεις μπορούν να εμφανιστούν και πολλά χρόνια μετά τη συνταξιοδότηση. Χρειαζόμαστε μια ολοκληρωμένη πρόληψη η οποία μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της συνεργασίας των επιχειρήσεων και των κρατικών αρχών στα κράτη-μέλη. Η αρχή της ε, προφύλαξης αποτελεί μια γενική αρχή της ενωσιακής νομοθεσίας. Δεν έχει ακόμη ξεκαθαριστεί ε, ε, σε ποιον βαθμό ε, η υγεία των εργαζομένων πλήττεται από τον χειρισμό τοξικών μειγμάτων. Και σε αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούν οι τροπολογίες που θα καταθέσω. Ευχαριστώ πολύ και σε εσάς, κύριε Αντελβού, λέει ο Πρόεδρος. Κύριε Λεπρετό. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα πω μερικά λόγια επί της αυτής. Είναι πολύ σημαντική. Πρέπει... να καταπολεμήσουμε τους... σε του καρκίνου. και να προσπαθήσουμε να καθορίσουμε τιμές οριακές για να αποφεύγονται παρόμοιες ασθένειες. Φυσικά συμφωνώ με τα όσα αναφέρονται στην έκθεση. Πιστεύω ότι επίσης θα πρέπει να κατατεθούν κάποιες τροπολογίες, διότι υπάρχει ένας τρόπος που παρουσιάζονται τα πράγματα που δεν είναι ο κατάλληλος. Είναι διότι όταν αναφέρεται ότι ο στόχος είναι να σώσουμε 100.000 ζωές μέχρι το 2069, εντάξει είναι σωστό σαν πρόθεση, αλλά αναφέρεται το εξής, κάτι που αποτελεί μια συνολική οικονομία από 34 έως 80 εκατομμύρια ευρώ. Ε, είναι δυστυχές αυτό, διότι είναι ατυχές, συγγνώμη. Διότι δίνουν την εντύπωση ότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι καταρχάς η οικονομία και εξοικονόμηση πόρων. Αλλά εμείς αυτό που θέλουμε να κάνουμε και να τονίσουμε είναι ότι θέλουμε να σώσουμε ζωές. Πρέπει λοιπόν να μην ε, ε, μας κατηγορήσουν ότι πέφτουμε στον τομέα του υλισμού. Ναι η Κομισιόν θέλει να πει κάτι επί του θέματος. Δεν βλέπω να έχει ζητήσει κάποιος από την Κομισιόν το λόγο. Να σας ενημερώσω ότι η προθεσμία κατά τροπολογιών είναι η 8η Δεκεμβρίου στις 12.00. Πρέπει να ξεπεράσουμε το σημείο 10 μοιραπουσιάζει η συγκίτρια. Περνάμε στα σημεία 12 και 13 που αφορούν ε, τον ε, εφαρμοστικό κανονισμό και κάποιες διατάξεις ε, σχετικά με τον κανονισμό 2007-2009 για, τα ευρωπαϊκά, για τα ενωσιακά σήματα και το ζήτημα της ε, κατάργησης της οδηγίας 2, μάλλον 95 και επίσης την οδηγία 216-96. Η κυρία Βίλκστρομ μας ενημέρωσε ότι δεν μπορεί να παραστεί διότι προεδρεύει στο πλαίσιο Επιτροπής Πέτη Αναφορών. Να δώσω λόγο στην Κομισιόν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να σας πενθυμίσω πολύ σύντομα ότι η βασική πράξη εδώ πέρα που έχουμε, ο κανονισμός δηλαδή, προβλέπει τη δυνατότητα τροποποίησης μέσω εκτελεστικών ή κατεξοδότηση πράξεων. Εμείς λοιπόν φασίσαμε να έχουμε έναν εκτελεστικό κανονισμό και έναν κατεξοδότηση κανονισμό και οι δύο έχουν συντηθεί στις πρώτες συνεδριάσεις που κάναμε το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο στα πλαίσια της δικής της Επιτροπής όταν συζητήσαμε τους εκτελεστικούς κανόνες και τους κατεξοδότηση κανόνες και συζητήθηκαν επίσης και στην ομάδα εμπειρογνωμών του Κοινοβουλίου όσον αφορά το νοσιακό σήμα. Τα κράτη-μέλη και εμπειρογνώμονες μας είπαν ότι ε, όντως βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο και αυτό επιβεβαιώθηκε και από τις δικές μάλλον και από τις ενώσεις ε, καταναλωτών, νέων και μέσω του, της ε, στο σελίδας που έχουμε στο διαδίκτυο. Και μέχρι τα τέλη λοιπόν του έτους και με τις συνεδριάσεις που προβλέπονται το Δεκέμβριο θεωρώ ότι θα μας σε θέση να οριστικοποιήσουμε τα δύο αυτά κείμενα. Θεωρώ λοιπόν ότι ε, βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο για την έγκριση των πράξεων αυτών τον Απρίλιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να μπορέσουμε στη συνέχεια να επεξεργαστούμε λίγο περισσότερο τον κατεξοδότηση κανονισμό. Εγκρίνοντα του δύο αυτού κανονισμού, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι για την βασική αυτή πράξη γίνεται μία τροποποίηση που θα έχει να κάνει με την αλλαγή τη αρρύθμιση που χρησιμοποιείται. Αναφέρομαι στο βασικό κανονισμό για το νοσιακό σήμα. Ήδη ξεκίνησε η διαδικασία αυτή στις 31 Οκτωβρίου και κινείται με την ταχύη διαδικασία μέσω των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρούμε λοιπόν ότι βρισκόμαστε σε καλό δρόμο, έχουμε προχωρήσει γρήγορα, θα καταφέρουμε να αντικαταστήσουμε όλους οι φυστάμενους κανόνες που πρέπει να αντικατασταθούν όσον αφορά το νοσιακό σήμα και θεωρώ ότι θα έχουμε καταφέρει αυτά μέχρι τις 31 Οκτωβρίου του 2017. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Ολοκληρώνονται και τα δύο αυτά σημεία, καθότι πιέζει πολύ ο χρόνος. Σας προτείνω να μην καλύψουμε τώρα το σημείο 11, το οποίο θα το κάλυπτε εγώ βασικά, και θα μπορέσω να σας ενημερώσω για την ερμηνεία και υλοποίηση της Οργανικής Συμφωνίας για τη Βελτίωση Νομοθεσίας αύριο το πρωί, όταν θα έχουμε και λίγο περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μας. Έχουμε τον κύριο Μπούντα μαζί μας, επομένω πάμε στο σημείο 25 εξέταση τροπολογιών όσον αφορά το συντονισμό συγκεκριμένων νομοθετικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων. Κύριε Μπούντε, έχετε το λόγο. Ας είστε σύντομος, παρακαλώ πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όντω, θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομο στην παρουσίαση αυτή. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι υπέβαλαν τροπολογίες, 193 ήταν συνολικά οι τροπολογίες, σημαντικός αριθμός. Συνάδελφοι από την Επιτροπή Γιούρι, και από άλλες επιτροπές υπέβαλαν τις τροπολογίες αυτές. Ελπίζω ότι οι συμβαστικέ τροπολογίε όντω θα αντικατοπτρίζουν την εργασία που έχουμε κάνει για το ζήτημα αυτό, προκειμένου να καταφέρουμε τελικά να έχουμε ένα τοπίο οπτικοακουστικών μέσων, το οποίο στην πράξη θα αντικατοπτρίζει όλες αυτές τις αλλαγές που βλέπουμε στο συγκεκριμένο κλάδο. Θα ήθελα απλώς να τονίσω κάποια σημεία που θεωρώ ότι είναι σημαντικά και τα οποία άπτονται της αρμοδιότητας της δικής μας Επιτροπής. Δεν μπορώ δυστυχώς να αποφανθώ για σημεία επί των οποίων αρμόδιες είναι άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές. Όλες λοιπόν οι τροπολογίες τονίζουν ε, ότι θα πρέπει να έχουμε μια ισορροπημένη προσέγγιση προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι αντικατοπτρίζονται όλες οι τεχνολογικές εξελίξεις, αλλά και ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού για όλους τους εμπλεκόμενους. Θεωρώ ότι ε, συμφωνούν οι περισσότεροι συνάδελφοι όταν λέω ότι θα πρέπει να έχουμε συνεκτικές και λογικές διατάξεις όσον αφορά τα νομοθετικά αυτά μέσα, προκειμένου να έχουμε από τη μία ανταγωνισμό και από την άλλη προστασία των καταναλωτών. Θέλουμε να διασφαλίσουμε την προστασία των καταναλωτών οι οποίοι χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες των οπτικοακουστικών μέσων, αλλά θέλουμε από την άλλη να διασφαλίσουμε και τα δικαιώματα του δημιουργού, το copyright. Θέλουμε να τονίσουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να παράγει κανείς ευρωπαϊκά έργα και να προωθεί κανείς τα ευρωπαϊκά έργα. Αυτός είναι ένα σημαντικός μας στόχος, γιατί η ευρωπαϊκή πολιτιστική πολυμορφία μπορεί να διατηρηθεί μόνο αν προστατεύουμε πραγματικά το copyright, τα πνευματικά δικαιώματα τα οποία συνδέονται με τα ευρωπαϊκά καλλιτεχνικά έργα. Και νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ισότιμη αμοιβή και όλων των συγγραφέων, καλλιτεχνών ή άλλων παραγόντων που παράγουν τα έργα αυτά. Ορισμένες τροπολογίες λένε ότι θα πρέπει να έχουμε ένα υψηλότερο επίπεδο προστασίας των ανηλίκων. Προφανώς το ζήτημα αυτό μας απασχολεί όλους. Όλοι θα θέλαμε να δούμε κοινού και συνεκτικούς κανόνες για όλους τους παρόχους ε, υπηρεσιών εκοκοστικών μέσων όσον αφορά την προστασία των παιδιών και των ανηλίκων ιδίω όσον αφορά το ψηφιακό εκείνο περιεχόμενο, το οποίο θα μπορούσε να πειράσει την διανοητική εξέλιξη των ανηλίκων. Πρέπει λοιπόν οι πάροχοι τέτοιων υπηρεσιών οπτικοκοστικών μέσων να δίνουν εκ των προτέρων επαρκείς πληροφορίες όσον αφορά το συγκεκριμένο αυτό οπτικοακουστικό περιεχόμενο. Επιθυμούμε επίση να τονίσουμε ότι θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να ταχθούμε κατά της πρόθεσης της ρητορικής μέσους, μίσους με συγχωρείτε, μέσω των οπτικοακουστικών μέσων. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν κάθε δυνατό μέσο προκειμένου τα οπτικοακουστικά μέσα και οι σχετικές υπηρεσίες σε εθνικό επίπεδο δεν θα πρέπει να περιέχουν, να περιέχουν καμία μορφή ρητορικής μίσους. Η έννοια αυτή της ρητορικής μίσους ξέρετε ότι καλύπτει πάρα πολλά πράγματα, από την τρομοκρατία μέχρι τον ρατσισμό ή την απλή εκδήλωση βίας, η οποία μπορεί να πάρει πολλές διαφορετικές μορφές. Επίσης, δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση στο πλαίσιο των υπηρεσιών αυτών να έχουμε φαινόμενα παρενόχλησης. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ιδίως όταν προσπαθούμε να προστατεύσουμε τους ανήλικους. Θέλουμε επίση και μέτρα πρόληψη τη ρητορική μίσου, όπω σα είπα, καθώ επίση και μέτρα πρόληψη του βίου περιεχομένου. Οι τροπολογίε λοιπόν που κατατέθηκαν τονίζουν ότι η ελευθερία τη έκφραση αποτελεί θεμελιώδε δικαίωμα, το οποίο δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί όμως ως μέσο απόκρυψης τέτοιων τοξικών πρακτικών. Είμαι στη διάθεση των συναδέλφων για περαιτέρω παρατηρήσεις και σας ευχαριστώ πολύ για τις τροπολογίες που καταθέσατε. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Δεν θέλει να πάρει κανεί το λόγο από ό,τι βλέπω. Δεν ξέρω αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να τοποθετηθεί για το ζήτημα αυτό, όχι. Μάλιστα. Πολύ γρήγορα. Λοιπόν, εξετάσαμε αυτές τις τροπολογίες, πρέπει να πω. Σημείο 25 ήταν αυτό και περνάμε στο σημείο 35 τα διάφορα. Εκεί υπάρχουν δύο θέματα και τον λόγο έχει ο κύριος Άντερσον για να μας τα παρουσιάσει. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εξέταση σχεδίου έκθεσης ή δύο σχεδίων, εκθέσεις, έκθεσης για την εφαρμογή της συνθήκης του Μαρακές. Όπως γνωρίζετε, πολλοί από εσά, η σύμβαση αυτή αφορά την πρόσβαση σε βιβλία, σε προσβάσιμη μορφής για τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης. 25 χώρες, Ινδία, Αυστραλία, Καναδάς, Βαζιλία, έχουν ήδη κυρώσει τη σύμβαση αυτή. Η συνθήκη έχει τεθεί σε ισχύ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως δεν έχει ούτε κυρώσει ούτε εφαρμόσει τη συγκεκριμένη συνθήκη. Και ένα από τα προβλήματα είναι ε, η κολυσιεργία στο Συμβούλιο που ελπίζω να ξεπεραστεί το συντομότερο δυνατό. Η Κομισιόν έχει προτείνει λοιπόν ένα κανονισμό και μια οδηγία που, αφορούν, που είναι και το αντικείμενο των δύο αυτών εκθέσεων. Πολύ σύντομα η Κομισιόν έχει παρουσιάσει πολύ καλές προτάσεις για την εφαρμογή της συνθήκης Φυσικά έχω και εγώ κάποιες τροπολογίες, 8 τον αριθμό, που ενισχύουν το μήνυμα και που εντάσσει στα κείμενα εφαρμογής τη διατύπωση που χρησιμοποιείται στην συνθήκη του Μαρακές. 25% ε, των τροπολογιών μου αφορούν και ορισμένε παραπομπέ στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών, ε, προσωπικών Δεδομένων. Πρόκειται για μια διαδικασία fast track προκειμένου να ασκηθεί πίεση στο Συμβούλιο ώστε το Συμβούλιο να αναλάβει επιτέλους δράση για τη συνθήκη του Μαρακές θα υπάρξουν γνωμοδοτήσεις από τις ε, Επιτροπές Απασχόλησης ε, και Πολιτισμού και στις 30 Ιανουαρίου θα διοργανωθεί και μια ακρόαση. Προθεσμία κατάθεση τροπολογιών είναι η 15η Δεκεμβρίου σύμφωνα με τις σημειώσεις μου και ψηφοφορία θα γίνει την 31η Ιανουαρίου. Μία από τις τροπολογίες θα ήθελα να σας παρουσιάσω, είναι και η σημαντικότερη, είναι η τροπολογία 2 για την οδηγία που αφορά την ενίσχυση του μηνύματος της ετολογικής σκέψης 11, όπου αναφέρεται ότι τα κράτη-μέλη δεν θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα επι, ε, ε, θέσπισης επιπλέον απαιτήσεων για την εφαρμογή της συνθήκης του Μαρακές. Εγώ με την τροπολογία μου αναφέρω ότι κάτι τέτοιο θα αντέβαινε τον, ε, τον σκοπό της συνθήκης και της οδηγίας. Το να θεσπίζονται γραφειοκρατικές διαδικασίες για την εκ των προτέρων επαλήθευση εκείνων που θα ε, διανύμουν ε, αυτά τα προσβάσιμα, ε, αυτές τις προσβάσιμες μορφές ε, είναι κάτι το οποίο θα καθιστούσε πρακτικά ανεφάρμοστη την ε, οδηγία. Γι' αυτό θεωρώ ότι η πρόταση Κομισιόν είναι καλή και η σημαντικότερη τροπολογία μου αφορά την ενίσχυση του μηνύματος ότι ε, πρόκειται για μια καλή πρόταση. Δεν πρέπει να υποσκάψουμε τη συνθήκη του Μαρακές καθιστώντας την, ανεφάρμοστη. Εμείς είμαστε ε, μια μεγάλη αγορά για ανθρώπους ε, ε, που αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης και για τα προϊόντα που απευθύνονται σε αυτούς. Ευχαριστώ πολύ, ο Πρόεδρος της Κομισιόν. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε πολύ σύντομα να σας πω. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσουμε τον κύριο Άντερσον και να ευχαριστήσουμε ευρύτερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τον δραστήριο ρόλο που έχει διαδραματίσει στην διαδικασία των διαπραγματεύσεων ε, της υπογραφής, της κύρωσης και της εφαρμογής της συνθήκης του Μαρακές. Είναι πολύ σημαντική η υποστήριξή σας προς εμάς και ε, είμαι βέβαιη ότι θα φτάσουμε γρήγορα στον, στον προορισμό μας, την κύρωση δηλαδή των εγγράφων αυτών, το συντομότερο δυνατό. Όπως είπε ο εισηγητής, εργαζόμαστε σε δύο μέτωπα. Πρώτον είναι η κύρωση της συνθήκης και δεύτερον η εφαρμογή της συνθήκης. Αυτό που συζητούμε σήμερα αφορά την εφαρμογή της συνθήκης, γιατί η κύρωση της συνθήκης, όπως γνωρίζετε, είναι ε, κάτι που η Κομισιόν έχει ήδη προτείνει στο Συμβούλιο τον Οκτώβριο του 2014. Δυστυχώς, ωστόσο, ε, βρίσκεται ακόμα στο στάδιο της συζήτησης για τη φύση των αρμοδιοτήτων και έχουμε ζητήσει απόφαση, γνωμοδότηση ε, του δικαστηρίου που ελπίζουμε να τη λάβουμε πολύ σύντομα. Πέραν του ζητήματος βεβαίως της κύρωσης πρέπει να συνεχίσουμε τη δουλειά μας όσον αφορά την εφαρμογή και αυτό είναι και το πακέτο που συζητούμε σήμερα. Μια διπλή νομοθετική πρόταση, οδηγία και κανονισμό, γιατί χρειαζόμαστε δύο διαφορετικά πράγματα. Πρώτον, να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει υποχρεωτική εξαίρεση στην εθνική νομοθεσία των κρατών μελών για, τους, ε, για τα άτομα με αναπηρίες και ταυτόχρονα τη δυνατότητα ανταλλαγής ε, ε, πληροφοριών για προϊόντα που απευθύνονται σε ανθρώπους με προβλήματα όρασης και αυτό είναι και η καινοτομία της συνθήκης, τον, τη δυνατότητα ανταλλαγής των μορφότυπων μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων κρατών που έχουν κυρώσει την συνθήκη. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να υπησέλθω σε λεπτομέρειες της πρότασης γιατί είναι σαφές ότι το Κοινοβούλιο ε, είναι ενήμερο. Απλά θα ήθελα να τονίσω ότι πρόκειται για μια πολύ συγκεκριμένη εξαίρεση. Πρόκειται για μια κλασική περίπτωση ε, αποτυχίας της αγοράς καθώς δεν υπάρχει αγορά εδώ πρόκειται για μια πολύ συγκεκριμένη και στοχευμένη εξαίρεση και γι' αυτόν τον λόγο η Κομισιόν θέλησε να διατηρήσει το πνεύμα της συνθήκης όπως ε, έτυχε της ε, μακροσκελούς διαπραγμάτευσης και θέλει να αποφύγει την επιβολή γραφειοκρατικών προϋποθέσεων που θα πλήξουν την πρόσβαση ε, των ανθρώπων με προβλήματα όρασης σε προϊόντα και σε μορφότυπα ανταλλαγής. Το Συμβούλιο επίσης ε, εργάζεται σκληρά υπό τη Σλοβακική Προεδρία και υπάρχει εύλογη ε, πρόοδος που έχει σημειωθεί. Έχουν συζητηθεί τα θέματα αυτά ήδη δύο φορές στην αντίστοιχη ομάδα εργασίας του Συμβουλίου επί των προτάσεων της Κομισιόν και ε, όπως είπα ε, έχουν συζητηθεί επί μακρόν. Προφανώς το Κοινοβούλιο αυτή τη στιγμή ασκεί ακόμη μεγαλύτερη πίεση ακολουθώντας πολύ ταχύες διαδικασίες, αλλά πιστεύουμε ότι αυτό μπορεί να βοηθήσει ως προς την ε, ταχεία ολοκλήρωση της διαδικασίας. Θα ήθελα λοιπόν για άλλη μια φορά να σας ευχαριστήσω και είμαστε στη διάθεση των βουλευτών για να συζητήσουμε ζητήματα που άπτονται των προτάσεών μας, όποιας φύσης και αν είναι αυτά, συμπεριλαμβανομένων των ζητημάτων τεχνικής φύσης και περιμένουμε με ανυπομονησία τις συζητήσεις που θα ακολουθήσουν το επόμενο διάστημα. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχει ζητήσει κάποιος τον λόγο για αυτό το θέμα, άρα μπορούμε να κλείσουμε το θέμα αυτό και θα συνεχίσουμε με συνεδρίαση και κλεισμένων των ε, θυρών των συντονιστών. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω από όσους δεν έχουν άδεια να παραμείνουν να εγκαταλείψουν την αίθουσα. Θα τα ξαναπούμε στις 6.30 για τη δεξίωση που διοργανώνει η Επιτροπή μας.